Σας καλώ λοιπόν να καθίσετε, λέει ξανά ο Πρόεδρος. Παρακαλώ καθίστε. Λοιπόν, ξεκινάει η συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση, νομίζω ότι η ημερήσια διάταξη είναι πλέον δεκτή. Γνωρίζω αγαπητοί συνάδελφοι ότι αρκετά μέλη της Επιτροπής μας δεν μπόρεσαν να είναι ανάμεσά μας σήμερα γιατί το αεροδρόμιο των Βρυξελών μόλις ουσιαστικά έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά του. Και αυτό μας οδηγεί άμεσα ξανά στην τραγωδία της 22ης Μαρτίου μια τρομοκρατικής ενέργειας και στο αεροδρόμιο αλλά και πολύ πιο κοντά μας στον πιο κοντινό σταθμό του μέτρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν χτυπήθηκε και ιδιαίτερα το Βέλγιο χτυπήθηκε. Νομίζω λοιπόν ότι από εδώ και πέρα εμείς θα πρέπει να ζούμε με αυτήν την τρομοκρατική απειλή. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να τελειοποιήσουμε τις συνεργασίες ανάμεσα στις αστυνομικές αρχές, τις αρχές συλλογής πληροφοριών και να αποδεχθούμε όλη την συστηματική ανταλλαγή των πληροφοριών που συλλέγονται για να μειώσουμε τους κινδύνους. Η σκέψη μας λοιπόν πάει στα τόσο πολλά δυστυχώς θύματα, 35 νεκροί και 300 τραυματίες χτυπηθήκαμε με ε, τρόπο και με βαρβαρότητα και γι' αυτό σας ζητώ ενός λεπτού σιγή ε, για τα θύματα και τις οικογένειές τους. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας μεταφέρω τώρα τις αποφάσεις τις οποίες κατέληξαν οι συντονιστές μας μόλις. Καταρχάς μια συμφωνία για την έκδοση μιας γνωμοδότησης Difference Initiative το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θέλησε να ορίσει τον εισηγητή, τον κύριο Γκονσάρες Πόνς. Ταυτόχρονα συμφωνήσαμε στην πρόταση Γκέιερ, μόνιμου εισηγητή μας για τις εξωτερικές υπηρεσίες, να ξεκινήσει μια μελέτη για το κόστος της απουσίας των εξωτερικών υπηρεσιών, δηλαδή τι θα κοστίσει στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν κάποιες από τις εξωτερικές υπηρεσίες αυτές δεν λειτουργούσαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μπορούμε εδώ να σκεφτούμε αν κάποιες τέτοιες υπηρεσίες δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να εξοικονομήσουν μερικές δαπάνες όταν θέτουν σε λειτουργία παράλληλα επικαλυπτόμενες εθνικές υπηρεσίες. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες, ο οποίος είναι ο ε, εισηγητής μας για τον προϋπολογισμό 2016 σχετικά με τον πρώτο διορθωτικό της χρονιάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή, αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού στόχο έχει να καλύψει την κατάσταση την έκτακτη αυτή που ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του άρθρου 172 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου ως προς τη νομική βάση και εδώ έχουμε και το είναι για τις το πρώτο διορθωτικό, το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού. Υπάρχει ένα μέσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες έκτακτες εφόσον υπάρχουν ανθρωπιστικές ανάγκες εντός των συνόρων μας είναι εργαλεία αυτά για να καλύψουμε ανάγκες και να βοηθήσουμε διαφορετικά από αυτά εκτός των σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι ακριβώς το εργαλείο για τις εσωτερικές ανάγκες, τις ανθρωπιστικές εσωτερικές ανάγκες. Το εργαλείο αυτό, το μέσο, δεν θα είναι προσωρινό για μια τριετία. Θα πρέπει να υπάρχει σε μόνιμη βάση και αν χρειάζεται, εφόσον χρειάζεται, να χρησιμοποιείται. Υπάρχει και το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ενεργοποιείται όταν υπάρχει κάποια φυσική καταστροφή. Και εδώ θα έχουμε αυτό το μέσο που θα ενεργοποιείται κάθε φορά που θα πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρειάζεται να αναλυθούν κάποιες δράσεις. Σε περιπτώσεις λοιπόν κατεπηγόντων, όπως συμβαίνει τώρα, θα πρέπει να ανταποκριθούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αυτό το σχέδιο δοτικού προπολογισμού με νέα πρόβλεψη για 80,2 εκατομμύρια ευρώ δέσμευση για πληρωμές Και ούτως ή άλλως συνολικά θα εκταμιευθούν 300 εκατομμύρια ευρώ για αυτές τις ανθρωπιστικές ανάγκες, τις έκτακτες ανθρωπιστικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 200 το 2017 και 200 το 2018 ένα σύνολο 700 εκατομμυρίων ευρώ αυτή την τριετία. Όλα αυτά βεβαίως έχουν να κάνουν με την κρίση των προσφύγων και για άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιδρά ανταποκρίνεται σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες, εφόσον απαιτείται δράση. Και εντός αυτού του πρώτου σχεδίου διευθυντικού προπολογισμού υπάρχει και ο στόχος να αναπτυχθούν οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Κεντρικού Καταπολέμησης της Δημοκρατία, εντός της Europol και οι αναγκαίες δεσμεύσεις για τις διάφορες δράσεις και τα 200 εκατομμύρια ευρώ που θα χρησιμοποιήσουμε από το Ταμείο για την ιστορική Ασφάλεια. Βεβαίως εγκρίνουμε αυτό τον διορθωτικό προπολογισμό δεδομένης της κατεπίγουσας ανάγκης. Απλώς θα απευθύνουμε κάποιες εκκλήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει καθ' όλη τη διάρκεια Τη διαδικασία, το νομικό πλαίσιο, όπως προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο για τον ε, προπολογισμό, προβλέπεται η συμμετοχή του Κοινοβουλίου και να αποφαίνεται το ίδιο. Ε, επίσης, λόγω του χαρακτήρα αυτών των κονδυλίων, του σκοπού που θα εξυπηρετήσουν, είναι ειδικά μέσα προφανώς, που θα πρέπει να παραμείνουν εντός των ορίων του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου και να συσχετιστούν να ενεργοποιούνται μάλλον, να χρησιμοποιούνται όποτε αυτό χρειάζεται μόνον θα εγκρίνουμε τα απαραίτητα περιθώρια από το, περιθώριο, από το περιθώριο των ε, κονδυλίων που δεν έχουν ε, δαπανηθεί 100 εκατομμύρια ευρώ από εκεί και είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε αυτή την έκτακτη ανάγκη οπότε πρέπει και να προβλεφθεί κάτι που φαινόταν προφανές η ανάγκη για να παρασκευθεί η ανθρωπιστική βοήθεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω ότι στο μέλλον αυτό το μέσο δεν θα διαρκεί μόνο τρία χρόνια, αλλά θα υπάρχει ώστε να χρησιμοποιείται όποτε παρίσταται ανάγκη. Η αλληλεγγύη κάποιες φορές επιδεικνύεται και με αυτόν τον τρόπο και αυτή τη στιγμή έχουμε μια κρίση που αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην πω όλη την ανθρωπότητα. Την κρίση των προσφύγων δηλαδή. Έχουμε υποχρέωση να βρούμε λύσεις. Γι' αυτό κάνω αυτή ακριβώ την πρόταση, για αυτό το σχέδιο διευθυντικού προπολογισμού, με αυτό το σχέδιο έκθεση, ώστε να υπάρξει κινητοποίηση, γοργή κινητοποίηση και εκταμείωση αυτή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λοιπόν. Είναι υπέρ ο Γενικός Εισηγητής. Είναι κάτι το οποίο εμπλέκει και τον προϋπολογισμό του 17 βέβαια. Ο κ. Γκάιερ, καταρχάς ευχαριστώ το Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες ο οποίος έχει καταθέσει μια έκθεση εξαιρετική. Είναι τόσο καλή που εμείς οι σοσιαλιστές δεν θα κάνουμε ούτε τροπολογία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και πόσο επιταχύνει τη διαδικασία. Όλα αυτά εγώ τα θεωρώ ε, υπεύθυνα από πλευράς δημοσιονομικής. Στους τρέχοντες προϋπολογισμούς έχουμε προβλέψει χρήματα ε, αρκετά για τους 160.000 πρόσφυγες που συμφώνησαν τα κράτη-μέλη ότι θα ε, κατανείμουν κανονικά. Συμφώνησαν θα το έκαναν αυτό και όφυλαν. Ε, να χρηματοδοτήσουν αυτή την επανεγκατάσταση. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν βαίνουν με την ταχύτητα που θα επιθυμούσαμε όλοι και που θα είχαμε φανταστεί. Άρα τα χρήματα αυτά δεν έχουν απορροφηθεί και ούτε πρόκειται να απορροφηθούν απολύτως το 2016. Γι' αυτό ε, είναι απολύτως ε, υπεύθυνο και σωστό αυτό που προτείνει ο Σοζέ Μανουέλ και θα έχει και αντίστοιχε επιπτώσει στον προπολογισμό του 2017. Δύο πράγματα. Ένα που θέλουμε να υποστηρίξουμε ρητά είναι το εξή. Στη συζήτηση που κάναμε ζήτησα μια νομική βάση ε, και δεν ξέρω αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσει, γιατί μου έλεγε πάντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποιο παράγραφο τη συνθήκη, αναφέρεται και βασίζεται για τι προτάσεις. Μα κανεί δεν αμφισβητεί τη νομική βάση και εγώ είμαι ο τελευταίο που θα το κάνω. Θεωρώ ότι είναι και επίγον και σημαντικό και χρήσιμο αυτό το εργαλείο και μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει την πρόταση και να οφείλει να το κάνει εγώ. Καθόλου αυτό δεν το αντικρούω, το αντίθετο, το καλωσορίζω. Πλην όμω πιστεύω ότι το μέσο αυτό, το εργαλείο, θα πρέπει να ε, έχει μια οδηγία για το πώς θα χρησιμοποιείται και να ορίζει και το Κοινοβούλιο πώς θα χρησιμοποιείται. Συμφωνώ με τον Φερνάντες. Δεν θα πρέπει τώρα να το συνδέσουμε για την αποδέσμευση των κονδυλίων με το συγκεκριμένο, ούτε ε, τροπολογία να κάνουμε, αλλά εγώ θα κάνω στα δικά μου κείμενα για τον προεπλογισμό του 2015 ε, την πρόταση ε, στο Κοινοβούλιο ότι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το νέο μέσο κάπως να το στοιχειοθετεί και κάπως να τακτοποιηθεί μέχρι τα τέλη του έτους μέσω οδηγίας για να δούμε την έγκριση, το στόχο, τα μέτρα που θα χρηματοδοτούνται, το πώς θα οριοθετείτε, την απαλλαγή. Υπάρχουν μια σειρά ζητημάτων ε, γιατί θα πρέπει να υπάρχει και διαφάνεια στη χρήση, θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό. Ένα δεύτερο που έχω και μια ερώτηση τεχνική προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ουσίας. Ε, λάβαμε την απόφαση ε, καταρχήν 160.000 πρόσφυγες να επαναγκατασταθούν. Και αν γνωρίζω και καλά, συμφωνήσαμε και με την Τουρκία, ε, ε, γίνεται λόγος για 72.000 Αυτό που συνδέεται 72.000 με τους 160 και το relocation. Οι 72 τώρα που είναι αντικείμενο της συζήτησης με την Τουρκία τι σχέση έχουν με τους 160.000, είναι τμήμα, είναι κλάσμα 72 ε, των 160 για την επανεγκατάσταση. Γιατί αυτούς που θα επαναπροωθούμε ε, μάλλον αυτούς που θα υποδεχόμαστε από την Τουρκία κάτι θα του κάνουμε, κάπω θα του υποδεχόμαστε, κάπου θα του εγκαταστήσουμε. Είναι 72 μέσα στου 160.000 ή πρέπει να προσθεθούν. Δεν το έχω καταλάβει και έχει και οικονομικέ και πολιτικέ συνέπειε. Δεν ξέρω, δεν το είδε κανένα άλλο, δεν μόνο εγώ έχω αυτή την απορία. Παρακαλώ, θα μπορούσατε να μου την απαντήσετε. Κύριε Κολμέλ, ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Γκάιερ. Συμφωνώ και ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τον κύριο Φερνάντες. Θεωρώ και εγώ ότι είναι εξαιρετική η έκθεσή του. Είναι απολύτως επίγουσα η κατάσταση και το αναγνωρίζει, αλλά ξεκαθαρίζει και κάποια θέματα αρχής που δεν θα πρέπει να είναι έτσι γενικά μετέωρα. Συμφωνώ απολύτως και υπογραμμίζω αυτό που είπε ο κύριος Γκάιερ, είναι σωστό πέρα από το γεγονός ότι θα πρέπει πολύ γρήγορα να απελευθερώσουμε κάποια κονδύλια για να βοηθήσουμε ορισμένους ανθρώπους, θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο βεβαίως να ξεκαθαρίσουμε τι κάνουμε και με ποιον τρόπο η βοήθεια αυτή θα υλοποιηθεί. Κύριε Γκάιε, δεν δηλώνετε μόνο εσείς άγνοια και εγώ την έχω αυτή την απορία και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, αλλά Ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να δημιουργήσουμε και τις συνθήκες εκείνες τις διαφάνειες που απαιτείται. Σήμερα αρχίζει ουσιαστικά η εφαρμογή της συμφωνίας με την Τουρκία και εγώ δεν έχω καταλάβει πού θα πάνε οι άνθρωποι αυτοί και πόσοι από την Τουρκία. Ε, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αλλιώς πάρα πολύ γρήγορα θα ζήσουμε καταστάσεις όπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίσουν άσκοπες και τέρμονες συζητήσεις. Από την αρχή λοιπόν να δούμε το θέμα αυτό ξεκάθαρα, να κάνουμε ένα λεπτομερές σχέδιο και να περιγράφονται εκεί και τα έξοδα, οι δαπάνες και τα λοιπά και ποια από τα έξοδα αυτά θα επιστρέφονται στα κράτη-μέλη. Τι κλίδα κατανομής έχουμε, τι τρόπο κατανομής και τι στόχους. Όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Πολύ καλή και ωραία η έκθεση, αλλά λείπει ένα μεγάλο ε, κεφάλαιο που έχει να κάνει με την υλοποίηση όλων αυτών. Ευχαριστώ, κύριο Μαραγά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ. Και θέλω να προσθέσω και τη δική μας στήριξη στην έκθεση του κύριου Φερνάντες. Είναι αναπόφευκτο να σκεφτούμε και τη συγκυρία και το γενικότερο περιβάλλον. Τώρα είναι οι μέρες που βγαίνουν όλες οι αμφιβολίες και οι αβεβαιότητες ή μάλλον οι αρνητικές βεβαιότητες ως προς την εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Επειδή είναι και κατεπήγον το θέμα και γενικότερα σημαντικό, αυτός ο διορθωτικός ε, και συμπληρωματικός ε, ε, προϋπολογισμός Ε, είναι ε, βεβαίως εκ των όνων Βεβαίως με την αίρεση ότι θα πρέπει να γίνει σωστή η εκτέλεσή του και υπεύθυνη. Δύο πράγματα να πω πάρα πολύ σύντομα. Πρώτον, για άλλη μια φορά, δεν ξέρω αν είναι νιωστή φορά που βλέπουμε πόσο είναι απαραίτητο να αναθεωρηθεί το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο όχι για να βάλουμε νέα ποσά και να συμπεριλάβουμε νέε δαπάνε, αλλά νέες ευθύνε, νέες δημοσιονομικές υποχρεώσει που έχουμε από τις νέες καταστάσεις που έχουν προκύψει. Αυτό είναι αναπόφευκτο, δεν πρέπει ε, να το αρνηθούμε. Το Κοινοβούλιο το ζητάει και θα πρέπει ε, απολύτως να αναθεωρηθεί το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο επιγόντως. Αυτό είναι πάγιο αίτημα της δικής μας Επιτροπής. Και ένα δεύτερο, μια ανησυχία που έχουμε για ε, τι θα γίνει με την υπηρεσία των οργανισμών για το άσυλο. Ε, μιλάμε για επανεγκατάσταση ε, για να Ε, Ξέρω ότι είναι τέτοια πράγματα που δεν μπορούμε να πάρουμε ε, άλλες αποφάσεις, αλλά ο Γραφείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας, το ΕΚΟ, αναλαμβάνει νέες ε, υποχρεώσεις. Θέλει πολύ έλεγχο όμως και προσοχή για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και εργαζόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Δεπρέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με όλους τους συναδέλφους. Θα συγχαρώ και εγώ τον εισηγητή μας, τον Χωζέ Μανουέλ, για την ποιότητα της εκθεσής του. Είναι μια έκθεση που καλύπτει όλες τις πτυχές που σε αυτή τη χρονική στιγμή πρέπει να ληφθούν υπόψη και να σχολιαστούν. Ήθελα να τονίσω καταρχά ένα στοιχείο που δεν είναι το πλέον σημαντικό από πλευρά προπολογισμού, όμω που παίρνει ιδιαίτερε διαστάσει στο σημερινό τοπίο. Δηλαδή οι ιδιαίτερε συνεισφορέ που απαιτούνται για την Europol και ιδιαίτερω για το κέντρο καταπολέμηση τη Τρομοκρατία, που άρχισε να λειτουργεί φέτο, στι αρχέ τη χρονιά, τα τραγικά γεγονότα στα οποία αναφερθήκατε πρόεδρε δείχνουν ακριβώ την καταπίκουσα ανάγκη που υπάρχει να ενισχυθεί συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με κοινέ δράσει ε, και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Το λέω και επιμένω ότι ε, τα δημοσιονομικά μέσα τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διατεθούν προ το κέντρο. Δεν βλέπω να υπάρχει αύξηση λοιπόν ε, στι δαπάνε, απλώ μετατόπιση. Να Εποφεληθώ, Πρόεδρε, για να συγχαρώ όλους τους και να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που έδειξαν την αλληλεγγύη τους προς το Βέλγιο και να παρατηρήσω ότι δυστυχώς αυτή η τραγωδία δεν αγγίζει μόνο το Βέλγιο. Ε, από τους 35 νεκρούς, 17 είναι οι Βέλγοι και οι υπόλοιποι είναι άλλων εθνικότητων και οι αναλογίες είναι παρόμοιες μεταξύ των τραυματιών. Άρα είναι μια τραγωδία που δεν έχει μόνο εθνικές διαστάσεις για το Βέλγιο, αλλά με τα διαφορετικές εθνικότητες των δικτύμων έχει ευρωπαϊκές και διεθνείς προεκτάσεις. Ε, όσο για τη δημιουργία αυτού του ταμείου ε, για τις κατεπήγουσες ανάγκες, τις έκτακτες ανάγκες, κατά την άποψή μου, Καλό είναι να διευκρινίσουμε το αντικείμενο, διότι δεν είναι πολύ σαφή εδώ τα πάντα. Κάποιες πιστώσεις απαιτούνται για την επαναγκατάσταση, όπως έχει ονομαστεί, το resettlement. Και κάποια δημοσιονομικά μέσα έχουν προβλεφθεί από το Ταμείο αυτό για από το αμύβ. Ε, μην μπερδέψουμε τα πράγματα λοιπόν. Δεν σημαίνει ότι 50.000. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν 50.000 άτομα που βρίσκονται μπλοκαρισμένοι στην Ελλάδα. Δεν θα γυρίσουν στην Τουρκία πριν από τις... γιατί είναι από... εκεί από τι αρχέ Μαρτίου. Και δεν ξέρουμε αν το θέλουν κιόλα. Ε, Προ στιγμή λοιπόν η κατάσταση αυτή είναι μάλλον επωνυδιστή, είναι δραματική. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αποκλεισμένοι στην ελληνική επικράτεια σε συνθήκε ε, πολύ κακέ. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η χειρονομία αλληλεγγύη και προ την Ελλάδα και αυτή η δημοσιονομική μα παρέμβαση για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την συγκεκριμένη κατάσταση, τη οποία δεν ξέρουμε ακόμα την έκβαση, την τελική έκβαση. Και δύο λόγια για τα αιτήματα που εκφράστηκαν, τι διάφορε εκκλήσει, γιατί είμαι μέλο και τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, Ελευθεριών του Πολίτη. Ο συνάδελφος ανέφερε ότι χρειάζεται μια συγκεκριμένη αξιολόγηση των, ε, ε, του αριθμού των ατόμων που θα πάνε προς την Τουρκία ή που θα έρθουν από την Τουρκία. Δεν μπορούμε όμως να το κάνουμε αυτό ακόμα. Δεν μπορούμε. Τι προβλέπετε να αποτρέψουμε όσο περισσότερο μπορούμε τους πρόσφυγες, οικονομικούς ή όχι, να φεύγουν από την Τουρκία για να πάνε στην Ελλάδα. Διότι όσοι ε, ε, από τις 20 Μαρτίου θα φύγουν από την Τουρκία για να πάνε στην Ελλάδα προβλέπεται να επαναπροωθηθούν προς την Τουρκία. Και οι Τούρκοι ήδη θα διώξουν κάποιου πρόσφυγε και μάλιστα και μερικού πρόσφυγε προ τα εσωτερικά τη χώρα. Οπότε δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι αριθμό θα φτάσει στην Τουρκία και θα προσπαθήσει από την Τουρκία να φύγει προ την Ελλάδα. Γιατί όλα εξαρτώνται από την λειτουργία τη συμφωνία. Και όσο περισσότεροι υποψήφοι πρόσφυγε υπάρχουν που θα φτάσουν ε, λαθρέα στην ελληνική επικράτεια και θα επαναπατριστούν στην Τουρκία, ε, τόσο περισσότερο κανόνας ένα προς ένα θα ισχύει και θα βλέπουμε κάποιοι πρόσφυγες που βρίσκονται ήδη στην Τουρκία επικράτεια να σπρώχνονται προς τα μέσα. Εδώ λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα τι αριθμός ανθρώπων θα έρθει. Είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο να προβλέψουμε ακριβώς τι θα συμβεί ε, και πώς θα διαμορφωθούν οι ροές. Με συγχωρείτε. Ε, μια παρατήρηση πρωτού ε, φτάσουν στην Τουρκία και επαναπροωθηθούν, θα καταγράφονται, θα καταγράφονται στα στοιχεία τους στην Ελλάδα. Και σε αυτή τη φάση μπορούμε να δούμε αν είναι οικονομική μετανάσταση... και αν του ξαναστείλουμε μέσα στην Τουρκία. Όχι όλους, όχι μόνο του οικονομικού. Ναι, για όλου. Ε, οι φάκελοι υποψηφιότητα για αιτήσει ασύλου θα καταγράφονται στην Ελλάδα. Ναι, θα καταγράφονται στην Ελλάδα. Με την παρουσία των εξωματικών συνδέσμων τη Τουρκία όμω. Αυτό προποθέτει ότι τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν διαθέσει ειδικού και συνεργάτε την Ελλάδα, στις ελληνικές αρχές, για να μπορούν να κάνουν τι καταγραφές. Ναι, γιατί για την ώρα τα πράγματα δεν έχουν πάει και πολύ καλά. Πολλοί από του υποψηφίου που έχουν φτάσει στην ελληνική επικράτεια δεν θέλουν να καταγραφούν τα στοιχεία του, διότι ξέρουν ότι θα του επαναπατρίσουν, θα του ε, επαναπροωθήσουν. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τι ροέ όσων έφτασαν πριν από τι 20 Μαρτίου και έχουν μπλοκαριστεί σε διαφορετικά σημεία, κυρίω στα σύνορα με τη Μακεδονία. Εδώ λοιπόν πρέπει ο μηχανισμό αυτό να αρχίσει να λειτουργεί, παρόλο που αυτό γίνεται με μεγάλη δυσκολία και για την ώρα τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Και υπάρχουν και φυσικά δυνέξεις μεταξύ των ομάδων μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν και αρ, αρκετά έντονες μεταξύ Σύρων και Πακιστανών, αρκετές συμπλοκές. Οπότε, εάν τα κράτη-μέλη δεν διαθέσουν ε, το, τους υπαλλήλους της Frontex που χρειάζονται και για την καταγραφή των στοιχείων και για τη διαχείριση των ε, επιχειρήσεων ε, υποδοχής και επαναπρόθεσης, η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Θα πάει προς το χειρότερο. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφωθεί στην πραγματικότητα. Ευχαριστούμε κύριε Κόλμελ. Θέλετε να ξαναπάρτε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα. Αγαπητέ συνάδελφε Ντεπρέ, δεν ξέρω, μήπως δεν εκφράστηκα αρκετά σαφώς όταν ζήτησα λεπτομέρειες. Φυσικά δεν ζητάω προγνωστικά εγώ τώρα ε, τι θα γίνει μέχρι τα τέλη του έτους ακριβή αριθμό, αλλά ειλικρινά τα όσα λέτε εσείς είναι εύγλωτη απόδειξη ότι χρειαζόμαστε περισσότερες λεπτομέρειες να γνωρίζουμε τώρα, να τις λύσουμε για να υπάρχει διαφάνεια. Δεν επιτρέπεται τώρα να έχουμε μια κατάσταση που θα πούμε ότι επειδή είναι δύσκολη η κατάσταση και δεν μπορούμε να αποφασίσουμε πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι όταν έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ποια χώρα δηλαδή. Πόσοι θα έρθουν, πού θα πάνε. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Bien. Monsieur... Καλώς. Ο κύριος... Ο έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ μετά τους υπόλοιπους συναδέλφους θέλω να συγχαρώ τον κύριο Φερνάντες για την εξαιρετική του έκθεση. Πέραν τούτου, να μου επιτρέψετε να κάνω ορισμένε παρατηρήσεις. Πρώτον, και εμείς είμαστε ιδιαίτερα διστακτικοί σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Το έχουμε επανειλημμένα πει. Άλλωστε, Θεωρούμε ότι η Ελλάδα δεν έχει τύχει της απαιτούμενης αλληλεγγύης και δημοσιονομικής στήριξης από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ευτυχώς, έστω και αν είναι κάτι το ανεπαρκές, ευτυχώς που κάποιες κατεπίγουσες λύσεις φαίνεται ότι αρχίζουν να βρίσκονται. Πέραν τούτου, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως έχει σήμερα σε εισαγωγικά βολεύεται με αναξιοπρεπή τρόπο. Η πρόκληση την οποία έχουμε απέναντί μας είναι πολύ μεγάλη πια και στην ουσία καλούμεθα εμείς να επικυρώσουμε κάποιες επιμέρους ρυθμίσεις οι οποίες δεν είναι ανάλογες με το μέγεθος της πρόκλησης που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε. Συνεπώς, ναι μεν υποστηρίζουμε τον συνάδελφο Φερνάντες για την καλή του έκθεση, αλλά αυτό δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση με μια σύμφωνη γνώμη της πολιτικής μου ομάδας για την αναξιοπρέπεια και ανηθικότητα αυτής της συμφωνίας για τους πρόσφυγες. Για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ επίσης και για τον λεπτό συγγύης που προηγήθηκε και το οποίο αποδεικνύει την λύπη και την ευαισθησία όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που εφήγησαν όπως και το Βέλγιο από τα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας. Σας ευχαριστώ επίσης που θα μπορέσω να δώσω κάποιες απαντήσεις στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Ξεκινώντας να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά το Κοινοβούλιο για την υποστήριξή σας, για την πρωτοβουλία, για την κατεπίγουσα βοήθεια προς τους πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν βρεθεί στην Ελλάδα και οι οποίοι είχαν ανάγκη από μια γρήγορη κινητοποίηση των δημοσιονομικών μέσων. Πρώτη ερώτηση, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Τέθηκε το ερώτημα και από τον κύριο Γκάιερ και τον κύριο Κολμέλ. Η λογική του ένας προς έναν, πού θα πάνε οι άνθρωποι αυτοί που θα έλθουν από την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος είναι καταρχάς οι 18.000 θέσεις οι οποίες υπάρχουν στην συμφωνία της 22ης Ιουλίου του Συμβουλίου. Υπήρξε μια πρώτη συμφωνία για το πού θα επανεγκατασταθούν τα πρόσωπα αυτά. 18.000 λοιπόν θα πάνε σε συγκεκριμένες χώρες μέλη ανάλογα με τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν οι χώρες αυτές. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μια τροπολογία στην απόφαση επανεγκατάστασης για άλλα 54.000 πρόσωπα επί τη βάση μιας εθελοντικής συμφωνίας. Στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να είμαστε λεπτομερέστεροι. Έχει προτείνει αυτή τη διεύρυνση του αριθμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα συζητηθεί αφού φτάσουμε στον αριθμό των 18.000 και αν υπάρξουν περισσότερες ανάγκες θα δούμε πώς θα τις αντιμετωπίσουμε μέσω μιας αντίστοιχης εθελοντικής συμφωνίας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο, από πού θα προέλθουν οι πιστώσεις. Εδώ θα ήθελα να διευκρινίσω το τι προτείνουμε. Καταρχάς, το Ταμείο για τους Πρόσφυγες. Εμείς δεν σημαίνει αυτό το οποίο προτείνουμε ότι δεν δίναμε βοήθεια κατεπήγουσα μέχρι τώρα αυτό που κάνουμε εδώ και αρκετό καιρό είναι να χρησιμοποιήσουμε τις πιστώσεις του ΑΜΙΦ που είχαν χρησιμοποιηθεί για κατεπίγουσα βοήθεια όλο όσο περισσότερο μπορούμε. Οι πιστώσεις αυτές δεν έχουν σαν στόχο αυτό που ονομάζουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν είναι δηλαδή χρήματα τα οποία είχαν ε, προσημειωθεί για να δοθούν για αγορά τροφίμων κτλ. Αλλά για άλλου είδους βοήθεια αλλά εμείς χρειαστήκαμε να τα χρησιμοποιήσουμε ε, και ένα σημαντικό ποσό πήγε στα κράτη-μέλη και στην Ελλάδα. Άκουσα ότι δεν έχει δοθεί βοήθεια στην Ελλάδα, έχει δοθεί σημαντικό ποσό, 180 εκατομμύρια ανάμεσα στο 15 και το 16 αυτή η κατεπίγουσα βοήθεια λοιπόν δόθηκε μέσω του άμυφ όσο αυτό ήταν δυνατό. Αυτό το οποίο πιστεύουμε είναι ότι αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια και αυτό το μέσο θα καλυφθεί επίσης και από τα 100 εκατομμύρια τα οποία δεν θα δαπανηθούν τους επόμενους μήνες θα μπορέσουμε να έχουμε επίσης γρήγορες μεταφορές στα στα διαφορετικά ταμεία και αν υπάρξει ανάγκη ενίσχυσης των ταμείων τότε θα απευθυνθούμε στις ε, επί των δημοσιονομικών αρχές. Πάντως βρισκόμαστε ε, σχετικά νωρίς στο 16 και δεν χρειάζεται να διαθέσουμε περαιτέρω ποσά εφόσον δεν έχουμε πλήρη εικόνα των αναγκών. Δεν ξέρω τι είπαν ακριβώς ο κύριος Μαραγκάλ και ο κύριος Ντεπρές. Στην ουσία αυτό το οποίο κάνουμε τώρα είναι μια χρήση των ποσών σταδιακή, ενδιάμεση, προσωρινή και προχωρώντας θα δούμε ακριβώς τι χρειάζεται να δαπανίσουμε για να αυξήσουμε, ε, ε, τις, να καλύψουμε μάλλον τις ανάγκες των τομέα της ασφάλειας και της μετανάστευσης. Λοιπόν, αυτά δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι. Όχι, ευχαριστώ πολύ, αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις σας. Θα έχουμε την δυνατότητα να επανέλθουμε στα θέματα αυτά. Νομίζω ότι θα αποδειχθεί τι δυνατότητες έχουμε να παίρνουμε τις αποφάσεις σε γρήγορο χρόνο. Γιατί αυτό έχει σημασία στην παρούσα περίπτωση να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών κατεπηγόντως. Η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι ένα σκάφος το οποίο είναι φτιαγμένο για τα γλυκά νερά μόνο. Νομίζω ότι και στην περίπτωση της Ελλάδας απεδείχθη πόσο κατεπήγον είναι το θέμα. Και εγώ θα συμφωνήσω λοιπόν με τα καλά λόγια που ακούστηκαν για τον κύριο Φερνάντες στις 11 Απριλίου θα ληφθεί η απόφαση, σε μία εβδομάδα δηλαδή στο Στρασβούργο. Και η έκθεση θα έρθει προς έγκριση στην Ολομέλεια του Στρασβούργου στις 13 Απριλίου. Έρχομαι τώρα στο μεθοριακό σώμα. Έπρεπε να το παρουσιάσει η κυρία Γκουαρτιά αλλά έχει προβλήματα μεταφορών για τους γνωστούς λόγους και γι' αυτό θα μας παρουσιάσει την έκθεση ο κύριος Γκάιερ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, επί το θέμα συνδέεται φυσικά με το προηγούμενο και έχει να κάνει με το εξή ζήτημα. Με ποιο τρόπο η Frontex θα μετεξελιχθεί σε έναν οργανισμό που θα αναλάβει περισσότερες ευθύνες στα ευρωπαϊκά σύνορα, τα εξωτερικά, επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή για τους πρόσφυγες και την προστασία των συνόρων είναι η Επιτροπή Ελευθεριών, ΛΥΜΠΕ, αλλά επειδή έχει και οικονομικό σκέλος, έχουμε και εμείς ε, το ρόλο μας και τη γνωμοδότησή μας. Την έχει εκπονήσει η συνάδελφος Γκάρδια Σάμπα. Οι τροπολογίες θα συζητηθούν στις 25 και 26 Απριλίου και θα αποφασιστούν εκεί. Η προθεσμία λύγει κανονικά αύριο το απόγευμα στις 6. Το θέμα δεν είναι τώρα η Frontex να γίνει ένας οργανισμός προστασίας εξωτερικών συνόρων που θα αναλάβει τη δουλειά αυτή από όλα τα άλλα αντίστοιχα που έχουν τα κράτη. Θα έχει ρόλο πιο υποστηρικτικό και πιο συντονιστικό σε σχέση με το σημερινό. Τα εξωτερικά σύνορα όπου αυτό χρειάζεται, όπου υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία, ιδιαίτερη επιβάρυνση για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημιουργηθούν εκεί pools, δηλαδή ομάδες προσωπικού από εθνικούς οργανισμούς και αρχές που θα υποστηρίζει και θα συντονίζει Frontex. Και προσωπικό που πολύ σύντομα μπορεί να συγκεντρώνεται και με υλικό, υλικό εξοπλισμό, αεροπλάνα, βαπόρια, αυτοκίνητα, οχήματα. Και θα πρέπει να δούμε εδώ εάν αυτό αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αν δηλαδή θα διευρυνθεί η λειτουργία της ε, Frontex, αν θα αυξηθεί το μέγεθός της και τι επιπτώσεις θα υπάρξουν. Η κυρία Γκαρδία Θαμπάλ έχει υποβάλει 11 τροπολογίες ε, για την πρόταση της, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ουσιαστικά αναφέρεται στους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν, στους εξωματικούς συνδέσμους, οι οποίοι θα αποσταλούν σε τρίτες χώρες και πώς θα εγκατασταθούν, πώς θα ενσωματωθούν στις αποστολές και τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλού. Και θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι εφόσον μιλούμε για οργανισμούς Και εφόσον η έδρα της Frontex βρίσκεται στη Βαρσοβία, δεν υπάρχει ακόμα μια επίσημη συμφωνία με τη χώρα υποδοχής της. Θα πρέπει αυτό κάποια στιγμή να λήξει. Διότι δεν είναι θέμα βεβαίως ευγένειας, είναι θέμα διοργάνωσης. Τι θα γίνει με τα παιδιά των υπαλλήλων της Frontex που εργάζονται στη Βαρσοβία λόγου χάρη. Υπάρχει και φυσικά μεγάλη σχέση με το κατά πόσον υπάρχει προθυμία. Βρίσκουμε ανθρώπους πρόθυμους να πάνε να εργαστούν εκεί. Θα πρέπει λοιπόν να επιληθεί το ζήτημα της έδρας και η πολωνική κυβέρνηση να καταλάβει ότι δεν μπορεί να παραμένει σε κρεμότητα το όλο ζήτημα για τόσο πολύ καιρό. Ε, εδώ πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια λύση και καθώς η Επιτροπή των Προπολογισμών και τα μέλη της ε, μπορούμε να αναλάβουμε δράση, καλό θα είναι να σκεφτούμε και την θέση του Γενικού Διευθυντή της Frontex, διότι αυτό προφανώς θα βρεθεί στο επίκεντρο των πολιτικών ε, συζητήσεων. Εάν ρίξουμε μια ματιά στις επιχειρησιακές ε, ευθύνες του Γενικού Διευθυντή της Frontex με τις νέες ε, προβλέψεις αυτές, εδώ προφανώς θα αυξηθούν αυτές. Δηλαδή δεν μιλάμε για γενικό διευθυντή του υπεύθυνου για τι επικίνδυνε χημικέ ουσίε, του οργανισμού αυτού τη Ευρωπαϊκή Ένωση που απλώ πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλα πηγαίνουν καλά και ότι συντονίζει τα πράγματα. Εδώ μιλάμε για παραβιάσεις δικαιωμάτων, την ευθύνη που μπορεί να του αναλογεί του ανθρώπου αυτού, την ε, συμπεριφορά των υπαλλήλων της Frontex κατά την ε, εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ο Γενικός Διευθυντής σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ε, απαιτείται να ασχοληθεί και με διαδικασίες επιπιθαρχικού εφόσον έχει υπάρξει κάποιο παράπτωμα ή κάποια παρατυπία. Νομίζω λοιπόν ότι η θέση αυτή του Γενικού Διευθυντή θα πρέπει να εγκρίνεται και από τα 28 κράτη-μέλη και θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλοι συμφωνούν και ξέρουμε ποια κριτήρια ισχύουν σε αυτές τις ε, περιπτώσεις. Εδώ πρέπει να λάβουμε λοιπόν υπόψη την πρόταση τη κυρία θα βάλει που λέει θα πρέπει να υπάρξει μια γραμμή στον προπολογισμό ώστε να καλύπτει αυτέ τι επιχειρησιακέ ευθύνε που θα αναλάβει η Frontex οι οποίε θα ε, γίνουν πολύ περισσότερε και να έχουμε και μια επισκόπηση για το πώ ε, χρησιμοποιούνται τα κονδύλια που διατίθενται για την εκτέλεση αυτών των ε, επιμέρου εξατομικευμένων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Frontex. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση της εκθέσεως Γουαρτιά Ζαμπάλ. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει το λόγο. Ο κ. Ντεπρέ. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Γκάιερ για την ευθύνη την οποία ανέλαβε να παρουσιάσει το έγγραφο αυτό των 82 άρθρων είναι σημαντικού μεγέθους και μάλιστα σε αυτή τη στρατηγική κατά τα άλλα στιγμή για τη σχέση του συντονισμού με τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Εγώ εξέτασα τις τροπολογίες που προτείνει η κυρία Γουαρία Ζαβάλ και συμφωνώ με τις περισσότερες από αυτές, αν και ίσως χρειάζονται και κάποιες άλλες για να γίνουν αρκετές αλλαγές και διευκρινήσεις κυρίως για τις ευθύνες της υπηρεσίας, ε, για τις αποσπάσεις ε, δυνάμεων και υπαλλήλων από τις χώρες μέλη και για τις συγκεκριμένες πλέον ευθύνες που αναλαμβάνει η υπηρεσία αυτή ε, και σε επίπεδο αστικής ευθύνης ακόμα. Ε, θα ήθελα τώρα να κάνω μια γενική παρατήρηση θα έλεγα για το Ευρωπαϊκό Σώμα Συνοριοφυλακών και Ακτοφυλακών. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ακριβώς το ότι δεν είμαστε σίγουροι όταν μιλάμε για τα σύνορα. Στο άρθρο 3 και στο άρθρο 5 τι λέγεται. Η Ευρωπαϊκή αυτή υπηρεσία, λέει το άρθρο 3, συνοριοφυλακών και ακτοφυλακών και τα κράτη-μέλη και οι υπηρεσίες των κρατών μελών στην ουσία εδώ μας δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει μία σύνοριοφυλακή ευρωπαϊκή και μία ακτοφυλακή ευρωπαϊκή ενώ από την άλλη είναι σαν να λέει ότι δεν υπάρχει αλλά υπάρχει σαν μορφή συντονισμού το άρθρο 5 τι λέει, η ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή αυτή εφαρμόζει τον ευρωπαϊκό τρόπο ελέγχου των σύνορων στα πλαίσια της κατανομής των ευθυνών ανάμεσα στα ευρωπαϊκά όργανα και στα εθνικά όργανα. Στην ουσία δίνουμε την ευρωπαϊκή ετικέτα και καθιστούμε υπεύθυνη την Ευρώπη για κάτι για το οποίο δεν είναι υπεύθυνη ή δεν είναι συνολικά υπεύθυνη, καθ' ολοκληρίαν υπεύθυνη. Αν διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο υπάρχουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία μετά από προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Frontex μπορεί να υποκαταστήσει τις εθνικές αρχές οι οποίες έχουν παραλείψει να κάνουν αυτά τα οποία καλούνται να κάνουν. Λοιπόν, είναι έτσι. Κοιτάξτε, είναι θέματα τα οποία δεν αφορούν συνολικά την πρόταση, αλλά με ενοχλεί συστηματικά να βάζουμε την ετικέτα της Ευρώπης πάνω σε τομείς τους οποίους η Ευρώπη δεν είναι πλήρως υπεύθυνη. Στα πλαίσια ιδιαίτερα ενός τόσο δηλητηριώδους κλίματος όπως το σημερινό. Αυτό δημιουργεί προβλήματα, σκεπτικισμό ε, σε πολλοί κόσμο. Γιατί ο κόσμος λέει ότι α, η Ευρώπη φυλάει πλέον τα σύνορα, παρόλα αυτά τα σύνορα τα διαπερνά οποιοδήποτε όποτε θέλει χωρίς έλεγχο. Κοιτάξτε πράγματι ανάμεσα στο κείμενο και στις προθέσεις ε, δυστυχώς και στην πραγματικότητα φοβάμαι ότι τα προβλήματα είναι δύσκολα. Με το PNR το ίδιο έχουμε. Θα υπάρξουν 28 PNR. Αν δεν σα είπα, λέει ο κ. Ντεπρέ, ότι είμαι υπέρ τη πρόταση. 300 εκατομμύρια κατέτος προβλέπονται εδώ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δαπανούν 30 δι το χρόνο. Για να καταλάβετε. Ο κύριος Μαραγκάη. Πρόεδρε. Εγώ θα συμμεριστώ το σκεπτικισμό του κυρίου Ντεπρέ. Νομίζω ότι ήδη μπορούμε να πούμε ότι το Frontex πρέπει να έρθει εδώ να μας εξηγήσει τι θα κάνει, πώς θα χρησιμοποιήσει τα μέσα αυτά, σε ποιους τομείς υπάρχει πλήρης ευρωπαϊκή ευθύνη και σε ποιους όχι. Δεν ξέρω πότε μπορεί να γίνει αυτό. Απαιτείται μια επαφή της Επιτροπής μας με τους υπεύθυνους του Frontex για να είμαστε πιο σωστά και λεπτομερέστερα ενημερωμένοι για την υπηρεσία αυτή η οποία μετατρέπεται σε κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Και να είμαστε βέβαιοι ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια υπηρεσία που θα ασχολείται με τις συλλογικές επαναπροωθήσεις και μόνον. ούτε και με μια υπηρεσία η οποία απλά θα κρατάει τους αριθμούς και τις στατιστικές αυτών που μπαίνουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό κινδυνεύει να γίνει. Βέβαια όλα αυτά δείχνουν ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είναι υπέρ της κατάργησης των εσωτερικών συνόρων, αλλά δεν εφαρμόζουν τη συμφωνία του Δουβλίνου, όπου η χώρα που θεωρείται υπεύθυνη είναι η χώρα στην οποία ο μετανάστης ε, πατάει για πρώτη φορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλήρης υποκρισία δηλαδή. Θέλουμε οι Τούρκοι να κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να γίνεται ε, από εμά. Ακόμα και αν γίνει κάτι τέτοιο στην Τουρκία, τότε θα ξαναρχίσουν να μπαίνουν από τη Λαμπεντούζα και την Ιταλία. Λοιπόν, κλείνει η συζήτηση παρακαλώ πάνω σε αυτό για την έκθεση Γκουατιά Ζάμπαλ, την οποία παρουσίασε ο κ. Γκάιερ. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Να θυμίσω ότι οι τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν πριν την 18η απογευματινή αύριο. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 26 Απριλίου και η επί της ουσίας έκθεση θα συζητηθεί τον Μάιο και στην Ολομέλεια η ψηφοφορία θα γίνει μετά το Μάιο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ερχόμαστε τώρα στις ψηφοφορίες. Σας ζητώ να βάλετε τις κάρτες σας στη μηχανή μπροστά σας. για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τον αριθμό των ψηφιζόντων. Λοιπόν, ξεκινάμε τις ψηφοφορίες. Έχουν μπει 20 κάρτες στο μηχάνημα. 12, 13 έχουν ψηφίσει μόνο. Ψηφίστε κάτι παρακαλώ. 16, 4 δεν έχουν ακόμα ψηφίσει δοκιμαστικά. 19 πλέον 21 ψηφίσαντες. Αλλά ένας δεν έχει ψηφίσει μάλλον. Λοιπόν τέλος της δοκιμαστικής. Η πρώτη έκθεση είναι το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Volvo Trucks, φορτηγά Volvo στην Ελβετία. Έκθεση Νεγκρέσκου. Τροπολογία υπαρίθμου 3. Ψηφίσατε όλοι. Ποιοι είναι υπέρ της τροπολογίας 3. Με προφορική τροπολογία διορθώνει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ για ανατάσσεως των χειρών. Κατά. Αποχές. Δεκτή η τροπολογία. Τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Με προφορική. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 6 άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας δεκτή τροπολογία 13 υπέρ 8 κατά Αυτά για την 6. 7 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 10 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 11 με προφορική του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή για το σύνολο του κειμένου τροπολογημένου πλέον Άρχεται η ψηφοφορία ονομαστική ψήφος. Πέρας της ψηφοφορίας 17 υπέρ, 4 κατά. Περνάμε τώρα. Περνάμε στην έκθεση Τη κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση για την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπή του συναδέλφου Νοβάκοφ. Ε, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. 11 προς 9 εγκρίνεται. 11 προς 9, ναι. Και μία αποχή. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 5. Πέρας. Εγκρίνεται 11 προς 9. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται 8 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται 9 υπέρ κατά Αποχέ, απορρίπτεται 10 υπέρ καλύπτεται και από την 9 οπότε δεν χρειάζεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 11 προς 9 και μια αποχή 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για το 14. πέρα. 11 προς 10 εγκρίνεται. Για το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικός άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται 16 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, μία αποχή. Τώρα, έλεγχος του Μητρώου των ομάδων εμπειρογνωμών της Επιτροπής. Η εισηγητριά μας, η κυρία Τρουιπέλ, θέλησε να αναβληθεί η ψηφοφορία αυτή, το ζήτησε. Και ο γενικό μα εισηγητή μα προτείνει κάποιε μεταφορέ. Του δίνω ευθύ αμέσω τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι μεταφορέ έχουν να κάνουν με τι εκθέσει που μόλι εγκρίναμε. Μεταφορά κονδυλίων στο 2 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Τα εγκρίναμε μόλις τώρα για του δικαιούχου στην Σουηδία, οι οποίοι απολύθηκαν, έμειναν άνεργοι στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανία. με 1.710.000 ευρώ και το άλλο είναι αυτό της τεχνικής βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με 380.000 ευρώ. Η άλλη έκθεση που εγκρίναμε δηλαδή. Ευχαριστούμε κύριε Γενική Εισηγητά. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Συμφωνείτε τις δύο μεταφορές θα τις ψηφίσουμε unblock μαζί. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Οπότε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Οι μεταφορές εγκρίνονται 12 προς 4. Δεν έχω άλλα ζητήματα στην ημερήσια διάταξη. Στα διάφορα. Έχετε κάτι να προτείνετε. Όχι. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι για τη συμμετοχή σας στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα λάβει χώρα στις 11 Απριλίου στο Στρασβούργο, στο τέλος του πρωινού. Πέρας της συνεδρίασης.